που αφορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δίνω το λόγο για ένα τετράλεπτο στην κυρία Μακοβέη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Μόλις συζητήσαμε την τρομοκρατία, είμαστε όλοι κατά της τρομοκρατίας. Η τρομοκρατία χρηματοδοτείται από την απάτη βασικά, από το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και η τρομοκρατία χρηματοδοτείται μέσω απατών κατά των ευρωπαϊκών ε, ταμείων. Μιλάμε για απάτες που ε, πλήττουν τα έσοδα και τα χρήματα των πολιτών. 3 με 5 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο αφορά η απάτη. Τεράστια αριθμή. Στην πραγματικότητα η κατάσταση θα μπορούσε να είναι ακόμα χειρότερη από αυτή που μας δείχνουν τα στοιχεία που διαθέτουμε και είναι απώλεια χρημάτων για τους νέους, για την απασχόληση, για την έρευνα, την καινοτομία. Μας κλέβουν τα λεφτά μας, μας κλέβουν τις ζωές μας, αυξάνεται η φτώχεια. Όλα αυτά λοιπόν ε, είναι συνέπεια, έχουν σαν συνέπεια ότι σήμερα δυστυχώς την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μάλλον οφείλονται στο ότι δεν έχουμε αποτελεσματικό μηχανισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να καταπολεμήσουμε την απάτη κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να πολεμηθούν οι απάτε κατά της Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό γίνεται από κάθε κράτο ξεχωριστά όμω σαν προσπάθεια και όχι συνολικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποια κράτη-μέλη είναι αποτελεσματικότερα στην καταπολέμηση των απατών αυτών. Άλλα κράτη-μέλη όμως δεν κινούνται καθόλου κατά των απατών ή είναι αναποτελεσματικά στην καταπολέμηση της απάτης αυτής. Υπάρχει διαφορά λοιπόν όσον αφορά την έρευνα των απατών ε, που στρέφονται κατά των συμφερών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Άρα χρειάζεται να έχουμε ενιαία υπηρεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο η οποία υπηρεσία να μπορεί να διεξάγει τις έρευνες όσον αφορά αυτού του είδους τις απάτες. Γι' αυτό είναι αναγκαίο να έχουμε ε, μια ευρωπαϊκή εισαγγελία, ένα κεντρικό φορέα. Οι απάτες έτσι θα καταπολεμούνται και θα ξυχνιάζονται πιο γρήγορα, θα γίνονται πιο γρήγορα οι έρευνες και η ανάκτηση των ποσών που εκλάπησαν θα είναι μεγαλύτερη. Θα αυξηθεί το ποσοστό ανάκτησης και σημαντικά πιστεύω. Να μην ξεχνάμε ότι εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα είμαστε οι θεματοφύλακες των χρημάτων. Είμαστε οι προστάτες των χρημάτων των πολιτών μας θα ήθελα αυτό το καθήκον να εκτελεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με τις διώξεις, έρευνες, έρευνες που στρέφονται κατά εκείνων που ε, υπάρχουν υπόνοιες ότι διαπράττουν αυτές πράξεις, να μπορεί λοιπόν τελικά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να προστατεύει καλύτερα το δημόσιο χρήμα. Χρειαζόμαστε Ευρωπαϊκή Υπηρεσία, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που να απαρτίζεται από εκπροσώπους ανεξαρτήτους, από εξειδικευμένους, από ειδικού εισαγγελείς, ε, να στραφεί κατά των απατών. Κάποιοι, εν μέρη οι εργασίες θα γίνονται ε, στα κράτη-μέλη και εν μέρη οι εργασίες θα γίνονται στο, στα κεντρικά γραφεία. Όλοι όμως αυτοί θα ανήκουν στην κεντρική υπηρεσία, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και θα συνεργάζονται. Μπορώ να κάνω μια σύγκριση. Η μόνη απάντηση είναι κεντρικό γραφείο, κεντρική υπηρεσία για την ε, καταπολέμηση απάτης. Αν καταπολεμούμε μια οργανωμένη ομάδα εγκληματιών που συστηματικά διαπράττει απάτες και μέσω πολλών κατών μελών, πώς μπορούμε να ανταποκριθούμε εμείς σε αυτού του είδους ε, το έγκλημα μόνο μέσω ε, μιας ε, ομάδας συγγελέων που θα παρτίζεται από μέλη όλων των κατών μελών και θα μπορούν να κινούνται γρήγορα και αποτελεσματικά αυτοί για να καταπολεμούν και να εξαλείψουν τελικά αυτό το μεγάλο πρόβλημα των απατών. Υπάρχουν ε, ερευνητικά μέσα. Κάθε φορά η έρευνα θα διεξάγεται σε κάθε κράτος μέλος με την άδεια του συγκεκριμένου κράτους μέλους με σεβασμό των ατομικών ε, δικαιωμάτων των υπόπτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Μακοβέη. Και τώρα το λόγο έχει η Επίτροπος, κυρία Γιωρόβα. Κυρίες και κύριοι αξιότιμοι βουλευτές, θα ήθελα να ξεκινήσω ε, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη μου προς την κυρία Μάκοβα και προς όλους τους κοιόδες συζητητές για την εντατική τους δουλειά στο θέμα αυτό. Αυτή η ενδιάμεση έκθεση παρουσιάζει την θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τον πιο σαφή δυνατό τρόπο. Και χαίρομαι ιδιαίτερω που υποστηρίζει τη γενικότερο στόχο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημιουργηθεί μια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η οποία θα είναι σε θέση να κάνει μια σημαντική διαφορά στην καταπολέμηση απάτη σε ό,τι αφορά τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Εγώ μέχρι το 2016 με, ε, προτίθεμαι να το θέσω αυτό σε λειτουργία για να δημιουργηθεί εισαγγελία και να υπάρξει σημαντική διαφορά σε ό,τι αφορά τα εγκλήματα κατά του προπολογισμού της Ένωσης. Ωστόσο, δεν το έχουμε πετύχει αυτό ακόμα. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται ακόμα στο Συμβούλιο και είναι πολύ περίπλοκες. Θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να εγγυηθούμε την ανεξαρτησία και την αποδοτικότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και θα ήθελα να αναφερθώ στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ως EPPO. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που υποστηρίζετε την ανοιχτή ε, διαδικασία διορισμού των μελών της Ευρωπαϊκής Εγγελίας. Επίσης, ε, συμφωνώ ότι χρειαζόμαστε σαφή καθορισμό των ε, εθνικών αρμοδιοτήτων και της Ευρωπαϊκής Εισηγγελίας και θα πρέπει να οργανωθεί η Ευρωπαϊκή Συγκυλία βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και οι διαδικασίες λειτουργίες θα πρέπει να συνάδουν με τις συνθήκες, με το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων και την Ευρωπαϊκή ε, Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Θα πρέπει να έχουμε ανεκτό μυαλό. Δεν υπάρχει κάποιο πρότυπο, δεν υπάρχει κάποιο προηγούμενο για την Ευρωπαϊκή Συγκυλία δεν υπάρχουν έτοιμες ε, λύσεις τις οποίες θα μπορούσαμε απλά να παράγουμε. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εξετάσει κατά πόσον το διασνοριακό καθεστώς ε, ερευνών θα πρέπει να ακολουθεί το μοντέλο που δίνεται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία ευρωπαϊκών ενταλμάτων. Αυτό το μοντέλο φαίνεται ότι δεν ενδείκνεται όμως για μια ευρωπαϊκή εισαγγελία γιατί πρέπει να λειτουργεί ως μια ενιαία υπηρεσία η ευρωπαϊκή εισαγγελία και θεωρούμε ότι η μεταφορά αρμοδιοτήτων για την δίωξη και την έρευνα περιπτώσεων απάτης θα πρέπει να έχει ένα sui generis καθεστώς για τις δυσυνοριακές έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σεβόμενο βέβαια το χαρτί των θεμελιωδών δικαιωμάτων και τις διαδικασίες. Θα πρέπει να γίνονται σεβαστές λειτουργικές ανάγκες και να ξεκινήσουμε από τα εργαλεία διακυβερνητικής συνεργασίας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τους λόγους άρνησης και το καθεστώς δικαστικής ε, αδειοδότησης, τους τομείς της δικαιοσύνης όπου θα δρά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ως ένα ενιαίο ευρωπαϊκό σώμα, δεν υπάρχει ανάγκη διπλής ε, εισαγγελικής αντιοδότησης και έγκρισης των ε, σχετικών μέτρων έρευνας. Θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να διασφαλίζει τις διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και αυτό θα απέφευγε το να επιβαρυνθεί υπερβολικά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, γιατί δεν μιλάμε για δεκάδες, μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες υποθέσεις κάθε χρόνο. Η συνθήκη επιτρέπει και μας καλεί να δημιουργήσουμε ένα συγκεκριμένο σύστημα το οποίο θα βασίζεται στην ιδιαίτερη φύση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αυτό που έχουμε προτείνει σέβεται τα δικαιώματα της αποτελεσματικής ε, δικαστικής αρχής και την ε, δικαιοδοσία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ως ε, εξοχήν όργανο ερμηνείας του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Σα ευχαριστώ, λέει πρόεδρο Και τώρα από την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων έχει ο κύριος Νεγκρέσκου το λόγο. Ευχαριστώ. Είναι πάρα πολύ θετικό το ότι έχει προχωρήσει αυτή η υπόθεση και εγώ είχα αναλάβει την γνωμοδότηση της Επιτροπής ε, της Νομικής για αυτή την έκθεση. Και έχουμε γνωμοδοτήσει και είπαμε ότι θα πρέπει ταχαίως να εγκριθεί αυτό το νομοθέτημα ώστε να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε την εγκληματικότητα. Όμως, ε, τρεις προτάσεις μας ε, δεν αντικατοπτρίζονται στο τελικό κείμενο. Πρώτα-πρώτα η ανεξαρτησία της αγγελίας ε, από τα πολιτικά κόμματα και όλων όσων ασχολούνται και σε εθνικό επίπεδο με την εισαγγελία και είπαμε επίσης ότι θα πρέπει να υπάρχουν εγγυήσεις για, ε, τη, για, τα φυσικά πρόσωπα που να παρέχονται την εισαγγελία και τρίτον ε, αρμοδιότητα κατά πολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος. Οπότε όλα αυτά όσον αφορά την ε, έκθεση που γιατί θεωρούμε ότι τελικά η εισαγγελία θα είναι, κάνει πιο αποτελεσματική θα πολέμηση του εγκλήματος. Τώρα, πολιτικές ομάδες. 1,5 λεπτό. Πρώτη κυρία Γκρέσλα. Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, η συζήτηση αυτή γίνεται για ένα σημαντικό θέμα και το πιο, σημαντικό πιο συνομιλητής απουσιάζει το Συμβούλιο, τα κρατη η Λιτωνική Προεδρία δεν έρχεται θα πάρει να συζητήσει μαζί μας για ένα θέμα το, για το οποίο το Συμβούλιο έχει αρμοδιότητα και όχι εμείς χάνει μια μοναδική ευκαιρία. Αυτά που έχουμε λοιπόν επιτάπητο για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν αρκεί ως πρόταση. Είναι καταδικασμένο σε αποτυχία και εμείς θα πρέπει να υπενθυμίσουμε στο Συμβούλιο ότι θέλουμε μια αποτελεσματική υπηρεσία. Δεν χρειαζόμαστε μια δυσκίνητη υπηρεσία και δεν, πρέπει να, και δεν μπορεί να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει, να καταπολεμάει, να καταπολεμάει δηλαδή τα διασυνοριακά εγκλήματα. Α, είμαι πολύ απογοητευμένη από το αποτέλεσμα και είμαι συνεισηγήτρια για το υλικό που έχει να κάνει με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πέντε τριμερείς διαλόγους έχουμε κάνει και προχωράει πάρα πολύ δύσκολο το θέμα αυτό με τα κράτη-μέλη. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια δυσκολία μεταφοράς αρμοδιοτήτων σε θέματα που έχουν να κάνουν με διακυβερνητική συνεργασία. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Συγγελίας για τις νοριακές περιπτώσεις φοροαπάτης, ε, όπου στην παρούσα φάση δεν ε, γίνεται σωστή δράση από τα κράτη-μέλη. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια δραματική κατάσταση για το θέμα τη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να καλέσουμε κάτι επιγόντω στο Συμβούλιο να μιλήσει μαζί μας. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρο. Μπλε κάρτα. Αποδέχεστε, κυρία Γκρέσλε. Δίνω λοιπόν το λόγο στην κυρία Φων Στόρκ. Κύριε Γκρέσλε, καλωσορίζω το γεγονός ότι αν σωστά κατάλαβα είσαστε κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελία, αλλά την καλωσορίζετε για διασυνοριακή εγκληματικότητα. Όντως έτσι είναι, για τη διασυνοριακή εγκληματικότητα πιστεύετε ότι χρειαζόμαστε ε, μια εισαγγελία εθνική για ένα κράτος που δεν υπάρχει, δεν είναι κράτος η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίσως θα πρέπει να μας εξηγήσετε λοιπόν αυτό. Ίσως κάτι να κατάλαβα κάτι λάθος. Πώς θα έχει δηλαδή εισαγγελέα η Ευρωπαϊκή Ένωση αφού δεν είναι κράτος. Κυρία Φωνστόρ, ξέρουμε ο, ποιος είναι το τομέας ειδικότητάς της Θα Ήθελα να σας πω ότι είμαστε υπέρ της εισαρχή νομική βάση στη συνθήκη της Λαβώνας ανεξάρτητα από ποια είναι η υποψή, ποια είναι η σας θα υπάρξει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ο Γενικός Εισαγγελέας μπορεί να εξετάζει διασυνοριακά εγκλήματα. Δεν χρειάζεται να υπάρχει κράτος. Η Πρόεδρος, ξέρω ότι ζητούνται α, και άλλες ε, μπλε κάρτες. Δεν χρειάζονται όμω πάντα μπλε κάρτε. Θέλω να είμαστε δίκαιοι. Για τρία λεπτά τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Κάφμαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε Επίτροπε το πόσο υψηλέ είναι οι ζημίε ει βάρος του ευρωπαϊκού προπολογισμού και οι ζημίε, δηλαδή ει βάρος και των ευρωπαίων φορολογουμένων κάθε χρόνο λόγω των περιπτώσεων απάτη, δεν το ξέρουμε ακριβώ. 500 ε, εκατομμύρια ευρώ, 2-3 δισεκατομμύρια, όλα αυτά είναι εκτιμήσει. Αυτό που ξέρουμε όμω είναι ότι η δίωξη ποινικών πράξεων από τα εθνικά κρατημέλη θα μπορούσε να είναι πολύ πολύ καλύτερη. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό δημιουργείται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ναι, όπως προβλέπεται και στη συνθήκη της Λισαβόνας και η κυρία Φωνστόρχια να βγάλει το διαβάσει άμα θέλει αυτά. Η εισαγγελία λοιπόν αυτή μπορεί, για προκειμένου τη εισαγγελία αυτή να μπορεί να αναλάβει τα καθήκοντά της κατά της, των, των περιπτώσεων απάτης κατά του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Η Ευρώπη λοιπόν μπορεί να δράσει και να πρέπει να μπορεί να δράσει για να προστατεύσει τα συμφέροντά τη και τα συμφέροντα των πολιτών της. Η ομάδα μας ε, υποστηρίζει λοιπόν επί της αρχής την ε, ίδρυση μιας Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Θα ήταν ένα σημαντικό βήμα για την σωστή προστασία των οικονομικών συμφέροντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ήταν ένα βήμα επίσης πάρα πολύ σημαντικό για την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Νομικού Χώρου. Τα κράτη-μέλη στην παρούσα φάση διαπραγματεύονται για τη διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και στη τελική ανάλυση θα πρέπει ομόφωνα να αποφασίσει το Συμβούλιο. Το Κοινοβούλιο δυστυχώ δεν συμμετέχει στην κανονική νομοθετική διαδικασία στο θέμα αυτό, αλλά το Συμβούλιο να ξέρει καλά, ακόμα και αν δεν είναι εδώ, ελπίζω να το μεταφέρει κάποιο το μήνυμα, να ξέρει λοιπόν το Συμβούλιο ότι θα πρέπει να συμφωνήσει και να εγκρίνει και το Κοινοβούλιο. Ε, ως εκ τούτου λοιπόν προκύπτει στη σωστή χρονική στιγμή η δεύτερη έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γιατί θεωρούμε, θεωρούμε ότι αποστέλει σαφή μηνύματα προς, τους, ε, το Συμβούλιο. Λευκή επιταγή δεν δίνουμε στα κράτη-μέλη. Θέλουμε καταρχάς ε, να υπάρχει ανεξάρτητη Ευρωπαϊκή Συγγελία, ανεξάρτητη από οποιαδήποτε περιοχή των κρατών μελών. Και εδώ πέρα χρειάζεται μόνο, όχι μόνο διαφάνεια, στη δράση των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, αλλά το Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετέχει στο διορισμό των ατόμων του Γενικού Εισαγγελέα. Θα χρειαζόμαστε επίσης διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων μεταξύ των ε, εθνικών αρχών και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά. Και εξίσου σημαντικό είναι οι κατηγορούμενοι και όσοι ευθύνονται για τέτοια εγκλήματα θα πρέπει να διώκονται σωστά. Επίσης δεν μπορεί να είναι μια δεύτερη δουλειά η δουλειά του Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να θέτουμε τις ε, αξιώσεις μας και θέλουμε να ληφθούν υπόψη αυτά από το Συμβούλιο γιατί ιδάλλως ε, θα εξαρτηθεί από αυτό μάλλον η έγκρισή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Κάφμαν. Έχουμε ένα έτοιμα για μπλε κάρτας και όπως σας είπα θα ακούμε έναν, μία μπλε κάρτα, να μιλητή. Θέλετε λοιπόν να αποδέχεστε την μπλε κάρτα. 30 δεύτερα κύριε Γιουρέκ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει συγκεκριμένο προϋπολογισμό, ίδιο προπολογισμό Πρόκειται περί πόρων, περί συνεισφορών των πολιτών και των κρατών μελών. Δεν φοβόσαστε ότι ο διαχωρισμός μεταξύ Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας από τις εισαγγελίες των κρατών μελών θα περιορίσει την αποτελεσματικότητα των αντιδράσεων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Μήπως είναι μια συγκέντρωση σε κεντρικό επίπεδο. Έχει 30 δευτερόλεπτα. Α, το αντίστροφο ισχύει, Στάνταλφε. Η εμπειρία μα δείχνει και δυστυχώ αυτό μα το είπε και η κυρία Μάκοβε, η συγγήτρια. Δυστυχώ ε, μία σειρά κρατών μελών δεν ερευνά αποτελεσματικά τι περιπτώσει αυτέ και έχουμε πολύ υψηλά ποσά απάτης. Γι' αυτό λοιπόν ξεκίνησε το έργο αυτό τη Ευρωπαϊκή Αγγελία και χαίρομαι ιδιαίτερω γιατί το πολέμησε το θέμα αυτό στην ε, συνέλευση την... Ε, με τη συνθήκη της Λισαβόνας για την καταπολέμηση της απάτης ακριβώς. Σας ευχαριστώ λέει πρόεδρος, επόμενος ομιλητής για ένα λεπτό, ο κύριος Κύρκοπ. Yes, thank you. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Επίτροπε, συμφωνούμε όλοι ότι η καταπολέμηση τη απάτη πρέπει να αποτελέσει πολιτική προτεραιότητα. Οι απάτε και η διαφθορά υπονομεύουν τη δημοκρατία μα και τι ελευθερίε. Όμω, πιστεύω ότι πρέπει να εστιαστούμε ε, επί εφαρμογής και διεύρυνσης των υπαρχών των εργαλείων. Olaf, Eurojust, Europol, EIO και, και η σχετική οδηγία που έχουμε. Δεν θα πρέπει να δίνουμε περισσότερα χρήματα και περισσότερους φόρους στην εθνική κυριαρχία. Ανταυτού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν ήδη αυτά που έχουμε. Αποτελεσματικό του τρόπο για να αντιταχθούμε στι απάτε είναι να σταματήσουμε να διαπράττει απάτη εν πρώτη όλοι συμφωνούμε από αυτού απλουστεύοντα τους κανόνες που διέπουν ε, του διάφορους τομεί του προπολογισμού της Ευρωπαϊκή Ενώσεω και βελτιώνοντας τον έλεγχο του προπολογισμού, αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος να πετύχουμε τους στόχους. Άλλη μια υπηρεσία, άλλη μια πολιτική γενική για ποικιλόμορφο πρόβλημα δεν είναι πραγματικά η βέλτιστη δυνατή λύση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κυρκό που δεχόσαστε γαλάζια κάρτα. Ο κύριος Γιάνκοβιτς. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Για πετε μας, κύριε, πώς θα ελεγχθούν αυτά οι πόροι, αυτά τα χρήματα. Γιατί και δεν λέω για τα κράτη-μέλη, λέω για τις άλλες χώρες. Λέμε για υποψήφιες χώρες. Αυτή μπορεί να γίνουν αποδέκτες ε, χρημάτων αλλά να μην τηρήσουν τα επισχυμένα. Εσείς κυρία Μακοβέη τι λέτε. Όποιος όμως ε, πληρώνει δεν θα μπορεί να έχει το δικαίωμα του να ελέγξει το πώς θα αξιοποιηθούν αυτά τα χρήματα γιατί θα αναλωθούν για το τίποτα. Κύριος Κύρκοπ, κοιτάξτε, είπα στα σχόλιά μου ότι είδαμε σημαντικό αριθμό υπηρεσιών διαθεσίμων εγώ θα ήμουν πρώτο να επικρίνω τις υπηρεσίες εκείνες. Τις επικρίνω τακτικά, διότι δεν θεωρώ ότι πάντα κάνουν τη δουλειά που τους ανετέθη. Βέβαια η προστασία των ευρωπαϊκών πόρων και χρημάτων έχει ε, προτεραιότητα. Αλλά δεν λέω ότι αυτή η συγκεκριμένη ιδέα και η νέα υπηρεσία θα κάνει πραγματική διαφορά όσον αφορά την ανάγκη και δυνατότητα των άλλων φορέων να εκπληρώσουν τις δικές υποχρεώσεις. Πιθανότατα λέγω. Ας συγκεντρωθούμε σε αυτά που έχουμε στα χέρια μας τώρα και ας τα βάλουμε να λειτουργεί σωστά. Ευχαριστώ για ένα δίλεπτο. Το λόγο έχει ο κύριος Μισελ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Λοιπόν, στην έκθεση αυτή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στέλνει ισχυρό μήνυμα προς το Συμβούλιο. Διότι ναι με ναι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αλλά όχι σε μια γραφειοκρατική δαπανηρή αναποτελεσματική δομή που εξαρτάται από τα κράτη-μέλη που κρύβονται πίσω από το θέμα της κυριαρχίας για να μην κάνουν τίποτα τα κράτη-μέλη κύριε Κυρκοπία. Κατά πολέμης απάτης είναι θέμα δεντολογικό για να εφαρμόζεται καλύτερο κράτος δικαίου και πρέπει να θέσει τέρμα στην κατάσταση ατιμορρησίας που επικρατεί πολύ συχνά η Ευρώπη πρέπει να επεξεργαστεί τα οικονομικά τη συμφέροντα χωρί να εξαρτάται την καλή θέληση των Ευρωπαϊκών Κρατών Μελών. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα επιτρέψει να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα τέτοιο μέσο. Κάποια κράτη-μέλη παίζουν διπλό παιχνίδι. Ε, το, στηρίζουν το μέτρο αυτό δημοσία, αλλά εκενώνουν από το περιεχόμενο αυτό το μέτρο και το αποδυναμώνουν ανεξάρτητη Ευρωπαϊκή Αγγελία θα δώσει πραγματική προστιθέμενη αξία και χαίρομαι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει στην έκθεση αυτή σειρά μέτρων συγκεκριμένων που ακολουθούν αυτή την κατεύθυνση. Η ανεξαρτησία μεταφράζεται βασικά, κυρία Κάφμαν, όπω το είπατε, από τη διαδικασία του καθορισμού των εισαγγελέων, από την κατανομή των αρμοδιοτήτων, δίνοντα προτεραιότητα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την δομή αυτή. Θα παρτίζεται από τμήματα που θα έχουν πολλούς ε, εισαγγελεί στο καθένα. Υπενθυμίζω, στο Συμβούλιο ότι η τελευταία κουβέντα την έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτό το θέμα και είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη η άποψη του Κοινοβουλίου μας. Ευχαριστώ. Κυρία Μισελ, υπάρχει γαλάζια κάρτα του κυρίου Ουγιαζόφσκι νομίζω. Παρόλο που δεν καθόστε σε σωστή θέση, νομίζω, άρα είναι δύσκολο για μας να βρούμε το όνομά σας. Κύριε Μισελ, καταρχάς δεχόσαστε τη γαλάζια κάρτα. Ευχαριστώ. Για 30 δευτερόλεπτα για την ερώτηση. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εξεπλάγην κάπως ακούγοντας τις παρεμβάσεις συμπεριλαμβανομένης αυτής του κυρίου Μισελ υπάρχει μεγάλη καχυποψία έναντι των κρατών μελών και των νομολογιών αυτών θα ήθελα να θέσω και το εξή ερώτημα με τη σειρά μου. Αυτός ο κανονισμός που αφορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μήπως θα μπορεί να επικυρωθεί ε, χωρίς την αποδοχή όλων των κρατών μελών ε, δυνάμει της συνθήκης. Αν είσαστε υπέρ μιας λύσης τόσο κεντρικής και με καχυποψία έναντι των κρατών μελών. Πρέπει να είμαι πολύ αυστηρή, λέει ο Πρόεδρος, λυπούμε λοιπόν, που σας διακόπτω. Δεν είμαι σίγουρος ότι πιάσα το πνεύμα της ερωτήσεως. Πρέπει να είμαι αυστηρός. Ε, κοιτάξτε, κύριε Πρόεδρε. Ε, ολοκληρώνω, ολοκληρώνω. Όχι, έχουν 30, όλοι έχουν 30 δευτερόλεπτα και το ξέρετε όταν ξεκινήσατε. Κύριε Μισελ, δεν ξέρω αν πιάσατε το πνεύμα της ερώτηση. Ε, έχετε όμω το δικαίωμα να απαντήσετε. Η ερώτηση, λέει ο κ. Μισελ, είναι κατά πόσο είμαι καχύποπτο έναντι των κρατών μελών. Είμαι καχύποπτο έναντι κάποιων κρατών μελών, σαφώ. Διότι ε, σειρά θεμάτων απατών πάντα ε, ε εκκρεμωδικούν στα κράτη-μέλη που πολύ συχνά παίζουν το χαρτί των συμφερόντων τους, του οράματός τους, της κυριαρχίας τους για να διαφύγουν ή να επιτρέψουν να ξεφεύγουν κάποιοι Οπότε επιβιώνει έτσι τιμωρησία. Γι' αυτό το λόγο είμαι για κεντρική αντιμετώπιση, για να υπάρχει νομολογία που θα είναι όλο και περισσότερο ενωτική, ενωμένη, ενιαία. Ευχαριστώ, συνάδελφοι, λέει Πρόεδρο. Ε, περνάει ο χρόνο, έχουν καθυστερήσει και έχουμε κανόνα 30 δευτερολέπτων για ερώτηση και απάντηση. Για ένα λεπτό, η κυρία Κάρη έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι απίστευτο το ότι η πρόταση που έχουμε διανύμει λέει ότι υπάρχουν 11 κράτη-μέλη που χρησιμοποίησαν την κίτρινη κάρτα διότι τα κοινοβούλια του θεωρούν ότι παραβιάστηκε η αρχή τη επικουρικότητας και ότι προχωρά το μέτρο πολύ μακριά. Αναφέρουν παραδείγματο χάρη ότι είναι δύσκολο για κάθε κράτος ε, μέλος να θέσει προτεραιότητες όσον αφορά το βάρος που δίδουν σε κάθε αδίκημα. Ε, θα πρέπει να θυμόμαστε εδώ ότι εδώ δεν μιλάμε μόνο για συνεργασία μεταξύ εισαγγελιών κρατών μελών, αλλά μιλάμε για ευρωπαϊκή εισαγγελία που θα έχει αποκλειστικές εξουσίες. Εδώ λοιπόν τα εθνικά κοινοβούλια ε, δεν ε, κάνουν επικρίσεις που δεν ευσταθούν. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να ξεπεράσει τα όρια ε, κάθε κράτους μέλους, του τι μπορεί να κάνει κάθε κράτους μέλος και η Εισαγγελία κάθε κράτους μέλους. Πρέπει να απορρίψουμε λοιπόν όλα αυτά. Ευχαριστώ ο κύριος Άλμπρεχτ, την επόμενος που έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχά, να ευχαριστήσω την κυρία Μακοβά, την εισηγήτρια, για τη σκληρή δουλειά που έκανα. Είναι σημαντικό το ότι έχουμε ένα αποτέλεσμα, μια διάμεση έκθεση, η οποία θα ε, προωθηθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, γιατί δεν είμαστε σε συναπόφαση από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ένα ναι ή ένα όχι, θα πούμε στο τέλο. Γι' αυτό λοιπόν είναι σαφές το μήνυμα. Τα κράτη-μέλη τα οποία δυστυχώ και πάλι δεν βρίσκονται εδώ στο, στην αίθουσα, αν δεν αποδεχτούν τίποτα από τις προθέσεις μας και από τις τροπολογίες που προτείνουμε, στην περίπτωση αυτή θα είναι αρνητική απάντηση σίγουρα για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θα πρέπει να το ξέρουν λοιπόν αυτό το κράτη-μέλη, αλλά είναι σαφές επίσης ότι εδώ στο Κοινοβούλιο μεγάλη πλειοψηφία εδώ και καιρό είναι υπέρ της δίδρυσης Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αλλά θα πρέπει να γίνει αυτό με τις σωστές συνθήκες, με τους σωστούς όρους και κυρίως να υπάρχουν οι σωστοί όροι λειτουργίας, αξιοπιστίας, διαφάνεια και θα πρέπει να είναι σαφές το τι ακριβώς θα πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει η Πρόεδρος. Μπλε κάρτα από την κυρία Φανστόρκ. Αποδέχεστε παρακαλώ την ερώτηση. 30 δεύτερα. Κύριε Άλμπρεχτ, καλωσορίζετε την εισαγωγή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας επειδή στα εθνικά κράτη-μέλη υπάρχουν προβλήματα απάτης και ε, σπατάλης ευρωπαϊκών πόρων. Όμως θα πρέπει να ιδρύσουμε μία νέα ευρωπαϊκή αρχή γιατί υπάρχουν προβλήματα σε μεμονωμένα κράτη-μέλη. Αυτό αποτελεί κατάφορη καταπάτηση της κυριαρχίας των κρατών μελών. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Άλμπρεχτ, έχετε 30 τεθρά για να απαντήσετε. Κύριε Φανστόρκη, νομίζω ότι κάθε απάντηση έχει να κάνει με την άγνοια της εξέλιξης του δικαίου. Φυσικά υπάρχουν ζητήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργηθεί από την κοινή ανάληψη της εθνικής κυριαρχίας διάφορων κρατών μελών. Κάποια θέματα λοιπόν τα κοιτάμε σε διεθνές επίπεδο ή μήπω θα αμφισβητήσετε και το Διεθνές Δικαστήριο με τη Διεθνή Εισαγγελία και πιστεύετε ότι αυτό αποτελεί ε, πρόβλημα και καταπάτηση της κυριαρχίας των κρατών μελών. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό τώρα κυρία Φερέρα. Ευχαριστώ πρόεδρε κύριε Φερέρα. τα πολέμηση της διαφοράς και του εγκλήματος και η προστασία των οικονομικών μας κοινότητας είναι κάτι ε, το οποίο είναι στην καρδιά του κινήματος των πέντε αστέρων. Οπότε γι' αυτό και θεωρούμε ότι είναι κάτι το θετικό να υπάρχει μια ανεξάρτητη εισαγγελία, ανεξάρτητη από τους πολιτικούς και έτσι να σταματήσουν οι ασυνέπειες, η αναποτελεσματικότητα και η ατιμορρησία που υπάρχει τώρα. Οπότε ε, θα πρέπει να θυμηθεί το Συμβούλιο του που δεν εδώ σήμερα ότι χρειάζεται μια καλή νομική βάση για να μπορεί να λειτουργήσει η εισαγγελία και γι' αυτό και ε, είναι πάρα πολύ θετικό και θα ήθελαμε μάλλον η οδηγία για την προστασία οικονομικής συμφερόντων να ε, τεθεί σε ισχύ σύντομα και να καλύψει και τα δικήματα σχετικά με τον ε, ΦΠΑ. Οπότε θα πρέπει να προστατευτούν έτσι τα οικονομικέ οικονομική ασφάλεια όπω όπως προβλέπει το άρθρο 86 της συνθήκης και όλες οι μαφίες και οι οργανωμένο έγκλημα να καταπολεμηθούν. Ο κύριος Φίλιππο, για ένα λεπτό. Κλασικά με μικρά βήματα θέλει να κάνει αυτή την, ε, ε, αυτή την πρόταση η Ευρωπαϊκή Τροπή και έτσι θα είναι κάτι που θα ξεπερνάει τα εθνικά δικαϊκά συστήματα θα αντικατασταθούν από αυτό το θεσμό. Οπότε θα πρέπει τώρα να έχουμε, λέει, η Επιτροπή ένα υπερ-εθνικό δίκαιο. Όμως το εθνικό δίκαιο είναι κάτι υπήρχε από την αρχαιότητα. Τώρα ο πολίτης θα είναι μόνος απέναντι ε, σε αυτό το θεσμό και έτσι δεν θα υπάρχει δημοκρατία ούτε θα γίνει τίποτα για τις εσωτερικές απειλές. Θα πρέπει όπως λένε οι αποφάσεις ε, των δικαστηρίων μας η δικαιοσύνη απονέμεται από τα γαλλικά δικαστήρια στη Γαλλία. Η εθνική δικαιοσύνη θα απέδιδε πολύ καλύτερα. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα είναι ένα γραφειοκρατικό τέρας, άχρηστο και αντιδημοκρατικό. Thank Έχετε μία μπλε κάρτα από τον κύριο Νεγκρέσκο. Την αποδέχεστε j'ai entendu euh, euh, votre prise de parole je dois vous dire que par exemple pour la roumanie et la bulgarie on a η Ρουμανία και η Βουλγαρία ωφελήθηκαν από την ανταλλαγή στοιχείων και από τη συνεργασία. Όμως η δικαιοσύνη δεν έχει χρώμα. Δεν θεωρείτε και εσείς ότι θα πρέπει να υπάρχει ευρωπαϊκή δικαιοσύνη. Εγώ δεν νομίζω ότι έχει πατρίδα η δικαιοσύνη. Όχι, νομίζω ότι η δικαιοσύνη, ακριβώς όπως και τα σύνορα, ο προπολογισμό, το νόμισμα, όπως και το δίκαιο, είναι τα βασικά χαρακτηριστικά ενός κράτους. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκός λαός. Πώς μπορεί να έχουμε ευρωπαϊκή δικαιοσύνη και υπερεθνικό δίκαιο. Δεν θα έπρεπε να έχουμε ε, ούτε, ούτε ευρωπαϊκό νόμισμα ούτε ευρωπαϊκό προπολισμό πάνω από τους εθνικούς και τα εθνικά νόμισμα. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν έτσι να αποσπάσουμε ε, τη δικαιοσύνη από την πραγματικότητα ενός ε, έθνους, ενός λαού. Αυτό, θα, αυτό είναι δικαιοσύνη. Για 1,5 λεπτό ο κύριος Σβέρ το λόγο. Ευχαριστώ. Καταρχάς να συγχαρώ την κυρία Μακοβέη για τη δουλειά που έκανε για το συγκεκριμένο αυτό θέμα. Νομίζω ότι είναι μια ιστορική απόφαση αυτή να συσταθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ακούσαμε πόσα χρήματα χάνονται, πόσα χρήματα χάνουμε εμείς και φορολογούμενοι κάθε χρόνο. Τα κράτη-μέλη δεν είναι αρκετά αποτελεσματικά όσον αφορά την ε, καταπολέμηση των απατών μόνο το 1 τρίτο των ε, αδικημάτων διώκονται πραγματικά και υπάρχει ανάκτηση των χρημάτων. Πρέπει να δημιουργήσουμε μια ανεξάρτητη εισαγγελία, ευρωπαϊκή εισαγγελία που είναι σε θέση να καταπολεμήσει το πρόβλημα. Και μόνο βάση ενός καθεστώτος sui generis θα μπορεί να είναι αποτελεσματικός ο φορέας αυτός. Εάν ε, ετοιμάσουμε άλλη μια χάρτινη τίγρη που θα βασίζεται μόνο επί συντονισμού, δεν θα αλλάξει τίποτα. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χρειάζεται νομιμότητα και θα λάβει νομιμότητα με την βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να υποδιαιρεθεί, να κατανεμηθεί το έργο της Όλαφ, της Europol και της Eurojust βάσει ενός συγκεκριμένου ε, νομικού πλαισίου για τα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Ευχαριστώ. Έχουμε γαλάζια κάρτα κύριε Σβέρ. Δέχεστε από τον κύριο Τσάνη γαλάζια κάρτα. Έχετε το λόγο κύριε Τσάνι. Yes, you have the floor, Mr. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Η ερώτησή μου είναι μια που ήθελα να απευθύνω στην κυρία Γκρέσσελα και εδώ ταιριάζει η ερώτησή μου. Μέχρι σότου έχουμε Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα έχουμε απάτες. Αν οι κυβερνήσεις των χωρών αν μια κυβέρνηση μιας χώρας αναμειγνύεται σε κάποια διαφθορά όπως με το Φίντες στη χώρα μου, μέχρι να έχουμε Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, πώς θα αντιμετωπίζετε αυτό το πρόβλημα. Ευχαριστώ η απάντηση σε 30 δευτερόλεπτα. Σας ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σαν υπηρεσία sui generis θα αποφεύγει τέτοιες περιπτώσεις όταν δεν αντιδρά σωστά ένα κράτος μέλος όταν ένας κράτος μέλος δεν καταπολεμά την ε, διαφθορά. 31% των συστάσεων της Όλαφ ε, ακολουθούνται από τα κράτη-μέλη. Μόνο 31%. Η ερώτηση είναι πόσες υποθέσεις ε, ολοκληρώνονται. Πιθανότατα λιγότερο από 31%. Χρειαζόμαστε συνεπώ με τέτοια υπηρεσία. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Για ένα λεπτό ο κύριος Νίτερ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Επιτροπέ, ένα από του προηγούμενου ομιλητέ είπε κάτι με το οποίο δεν συμφωνώ. Γιατί πιστεύω ότι χρειάζεται κατεπηγόντω η ευρωπαϊκή εισαγγελία. Ιδιαίτερα επειδή σε κάποια κράτη-μέλη υπάρχουν σημαντικά προβλήματα σε ό,τι αφορά του ευρωπαϊκού πόρου που κατασπαταλώνται, ε, υπεξαιρούνται και όλη αυτή η διαφθορά υπονομεύει ασφαλώς την εμπιστοσύνη των πολιτών και των ε, εκλογέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί βλέπουν, δεν βλέπουν πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση τους βοηθάει, πώς τους βοηθάει να πετύχουν τους στόχους τους. Χρειαζόμαστε λοιπόν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εντελώς ανεξάρτητη από τα κρατημέλη, γιατί γνωρίζουμε ότι υπάρχουν διάφορα κρατημέλη τα οποία δεν θα θέλουν να τηρήσουν τους συμφωνημένους κανόνες και να καταπολεμήσουν τη διαφθορά. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται κατεπηγόντως αυτή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ευχαριστώ κυρία Στίβενς για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αξιότιμοι συνάδελφοι, είμαστε, είμαι υπέρ ε, της καταπολέμησης, ε, της κατασπατάλησης και της επεξαίρεσης ευρωπαϊκών πόρων. Αυτό δεν σημαίνει ότι η ίδρυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ως ανεξάρτητη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία αποτελεί τη σωστή λύση. Έχουμε ήδη τη Eurojust για την δικαστική συνεργασία και την Ολαφ που είναι αρμόδια υπηρεσία για την καταπολέμηση της διοικητικής απάτης. Με άλλα λόγια, το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί σε άλλο επίπεδο πιο αποτελεσματικά γιατί ουσιαστικά η ίδρυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποτελεί ουσιαστικά κατασπατάληση των ευρωπαϊκών πόρων. Το άρθρο 86 α, της συνθήκης αναφέρει ότι θα πρέπει η ευρωπαϊκή αυτή αρμοδιότητα να προέρχεται και να μείνει στα χέρια των ήδη υπηρεσιών και της Eurojust. Βρισκόμαστε επίση σε φάση τριμερούς διαλόγου ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Γι' αυτό λοιπόν είναι λανθασμένη αυτή η χρονική συγκυρία για την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Χρειάζονται κάποιε συστάσει και θα πρέπει επίσης το Συμβούλιο τελικά να έχει και τη δική μα έγκριση. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Our next speaker for one and... Ευχαριστώ. Ένα μισή λεπτό τώρα το λόγο έχει ο κύριος Dartmouth. Uh, just yesterday... Μόλις χθες ο Γάλλος πρόεδρος εξέφρασε την κριτική του κατά προβουλευτούν. Είπε ότι η Γαλλία ποτέ δεν θα εγκρίνει καμία τροποποίηση όσον αυτό το θέμα. Και φαίνεται ότι τελικά το πακέτο αυτό τελικά θα σταματήσει αυτή η σπατάλη με το Στασβούργο. Και φαίνεται ότι αυτή η σπατάλη είναι ένα, κάτι που ταιριάζει και με το θέμα του Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Αλλά δεν θα συμβεί αυτό ποτέ. Ο πρόεδρος της Γαλλίας μπορεί να είναι επικριτικός όπως πάντα. Επίσης επικρίνει τη δημοκρατία η έκθεση. Αυτοί που συνέταξαν συνθήκες της Αβώνας γνωρίζαν πολύ καλά ότι μια πρόταση για Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα ήταν κάτι απαράδεκτο για τις εθνικές κυβερνήσεις και πράγματι 14 εθνικά κοινοβούλιο ε, πρόβαλαν βέτο αλλά έχει εισαχθεί μια ρήτρα ντροπή κιόλας ούτω ώστε τα κράτη-μέλη θα μπορούν μέσω διευρυμένη συνεργασίας να προχωρήσουν όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είναι αξιόμεμπτο αυτό, όμως η έκθεση μας υπενθυμίζει το θέμα της διαφθοράς και της απάτης κατά των πόρων τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Πάνω από τρία δις το χρόνο κλέπτονται. Τι δείχνει αυτό, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλογεί σε κάποιο είδος παρασίτου τρέφεται η Ευρωπαϊκή Ένωση από τον φορολογούμενο. Και όπως λέει η έκθεση, τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τροφοδοτούν το κόστος τη εσωτερική διαφθορά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι δούριο ύπο αυτή η πρόταση, δεν λύνει τίποτα. Καταστρέφει ακόμα περισσότερο την εθνική κυριαρχία. Χώσαστε γαλάζια κάρτα. Η κυρία για 30 δευτερόλεπτα. Είσαστε διατεθειμένοι να σημειώσετε ότι ο Γάλλος Πρόεδρος προασπίζει το ευρωπαϊκό δίκαιο που κατοχυρώνεται στις συνθήκες και που έχει να κάνει με την σημερινή διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Um, Απάντηση. Κοιτάξτε. Ήταν κομψή η ερώτηση βέβαια αλλά εγώ γιατί διαμαρτύρομαι και το κόμμα μου ότι το ευρωπαϊκό δίκαιο υπερτερεί του, ε, ε, του κοινού δικαίου της Βρετανίας, του Common Law, που είναι πολύ ανώτερο σύστημα. Όποιος είναι σοβαρός όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και άνθρωποι σαν και εσάς είσαστε σοβαροί, εγώ δεν είμαι, πιστεύω ότι είναι σπατάλη χρημάτων και χρόνου είναι απίστευτο ότι ε, υποστηρίζετε τον πρόεδρο της Γαλλίας και υποστηρίζετε αυτό το να ερχόμαστε στο Στρασβούργο 12 φορέ το χρόνο. 30 δευτερόλεπτα έχετε, λέει η Πρόεδρο. Προσπαθούμε να είμαστε πολύ δημοκρατικοί και να δίνουμε σε όλου το λόγο. Ευχαριστώ λοιπόν. Επόμενο για ένα λεπτό η κυρία Μάιερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, πληρώνουμε κατά εντολή των Βρυξελών και εξοικονομούμε την εντολή των Βρυξελών και σε λίγο θα κάνουμε και δίωξη την εντολή των Βρυξελών. Ευρωπαϊκή σημαία, ευρωπαϊκό α, ύμνο, ευρωπαϊκή εισαγγελία, η Ολλανδία και 10 άλλες 10 ε, χώρες βγάλαν κίτρινη χάρτα και τους ε, μουτζώσαν ουσιαστικά. Είμαστε κατά τη διεύρυνση αρμοδιοτήτων, όχι μόνο για τη δίωξη τη απάτη, αλλά και για την τρομοκρατία, την ε, απαγωγή ε, παιδιών και ένα σωρό άλλε αρμοδιότητες θα χρειαστεί στο μέλλον να τι δώσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχει τίποτα να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ η Ευρώπη. Πρόκειται όχι για δίωξη απάτη, αλλά για εξουσία. Δεν υπάρχει περιθώριο για τα ναζιστικά κράτη. Ελπίζω αυτό να το έχουν υπόψη οι συνάδελφοι αύριο που θα ψηφίσουν. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό τώρα το λόγο έχει η κυρία Τσινίτση. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Πρόκειται για την πιο φιλόδοξη ε, προοπτική που έχουμε όσον αφορά αυτό το θεσμό της ε, ε, εισαγγελίας. Ευχαριστούμε την κυρία Μακοβέ. Θα πρέπει να ακουστεί η φωνή του Κοινοβουλίου να περάσουμε αυτά τα όρια, τα όρια που θα πρέπει να αποτελούν την περιχαράκωση του τι θα πρέπει να εγγυηθεί τη λειτουργία αυτής της αγγελίας θα πρέπει να υπάρχει ανεξαρτησία από τα κράτη-μέλη και από τα θεσμικά όργανα. συνεργασία αποτελεσματική με τα κράτη-μέλη, αποτελεσματικοί μηχανισμοί για έρευνα και για συλλογή των αποδείξεων και τελευταίο αλλά σημαντικό θα πρέπει να υπάρχει σε κάθε φάση της, σε κάθε φάση της οικονομική να υπάρχει σεβασμός των δικαιωμάτων των ε, κατηγορουμένων. Ο κύριος Ένα λεπτό. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αυτό το είπαμε, το είπε και ο κύριος Μισελ να σεβαστούμε τις νομικές παραδόσεις του κάθε κράτους μέλους. Δεν συμφωνώ με την έκθεση Μακοβέη, δεν μπορώ να την ψηφίσω, γιατί αντιβαίνει σε όλα αυτά που σας προανέφερα. Εννέα κράτη-μέλη έδειξαν την κίτρινη κάρτα. Δεν θέλουν Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Χρειάζεται ομοφωνία για να συγκροτηθεί αυτή η εισαγγελία. Για αυτό και αυτό το οποίο θα προκύψει θα είναι κεντροκατευθυνόμενο, ανώτερο των κρατών μελών. Θα έχει ταυτόχρονα σαν αρμοδιότητα καταπολέμηση της απάτης, αλλά και την καταπολέμηση του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος. Να τι θα η δεύτερη φάση για τη συγκρότηση μιας τέτοιας αγγελίας. Θέλετε να διευρυνθούν οι αρμοδιότητες, αλλά τελικά η εισαγγελία θα είναι ανύπαρκτη, γιατί θα είναι πάρα πολύ κεντροκατευθυνμένη. Ένα λεπτό κύριε Ρέγνερ. Πρόεδρε, εδώ και 10 χρόνια και παραπάνω μιλάμε για την ανάγκη Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και θα ήθελα στο απόν Συμβούλιο να υποθυμίσω την περίφημη υπόθεση ε, για, το Ευρωπαϊ... για το ελληνικό καλαμπόκι. Εδώ το Ευρωπαϊκό Δικαστόριο... Δικαστήριο αναγνώρισε την ανάγκη προστασίας ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο των ευρωπαϊκών συμφερόντων στο ίδιο επίπεδο όπως τα εθνικά συμφέροντα. Είναι μια λογική λοιπόν μεταξέλεξη αυτής της αρχής η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Υποστηρίζω λοιπόν απόλυτα τον στόχο προστασίας των ευρωπαϊκών συμφερόντων και την καταπολέμηση της απάτη. Και πιστεύω ότι είναι λογικό αυτό για όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου. Θα ήθελα όσους ε, αμφιβάλλουν εδώ στην αίθουσα να τους επενθυμίσω τη συνθήκη της Λισαβόνας που τονίζει την καταπολέμηση βαρέων ποινικών ε, αντικειμάτων στο θέμα του προπολογισμού και τη κατασπατάληση πόρων. Και θα ήθελα να πω ότι η κυρία Μάκοβε έκανε σπουδαία δουλειά. Ευχαριστώ, κύριο Γιούρεπ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Για το θέμα τη Ευρωπαϊκή Αγγελία πρέπει να πούμε ότι τα κράτη-μέλη, τα κράτη, ε, τα έθνη κράτη είναι το θεμέλιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Δεν μπορούμε να το αμφισβητούμε αυτό, διότι αμφισβητούμε από την ε, συνεργασία μας και θα στερηθούμε συμβαλόμενα μέρη. Άλλαξε με να αλλάζει το χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αρχή. Το κοινό νόμισμα ήταν το εργαλείο και το μέσο ε, του εμπορίου και τώρα γίνεται το ενιαίο νόμισμα ένα εργαλείο δημοσιονομικό. Το ίδιο ισχύει και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η προλαλήσα σας συνάδελφος ανέφερε το άρθρο 86 της ε, συνθήκης αλλά το άρθρο 4 προβλέπει, στην ίδια συνθήκη το άρθρο 4 προβλέπει την επέκταση των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής ε, Εισαγγελίας. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να έχει πολλά κοινά συμφέροντα δεν μπορούμε να προχωρήσουμε καταστρέφοντας τα θεμέλια μας, δημιουργώντας πολλούς κοινούς ε, θεσμούς. Τώρα είμαστε στο Catch the Eye, έχουμε πέντε αγορητές, για ένα λεπτό. Ο κύριος Βος έχει το λόγο. Vielen Dank. Ευχαριστώ. Καταρχά, θα ήθελα να επιβεβαιώσω για μία φορά ακόμα ότι η εισαγωγή μια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι σημαντική. Και γι' αυτό λοιπόν θα το προωθήσουμε. Εγώ θα ήθελα στο πλαίσιο αυτό να είχαμε μία συνολική ιδέα. Και όχι μόνο να υπήρχε μία Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά πέραν αυτού να υπήρχαν και οι δομές που χρειάζονται τι θα συμβεί για παράδειγμα με τη Eurojust, πώς θα δημορφωθεί η κατάσταση, υπάρχουν ε, και προτάσεις τι θα γίνει με τη Europol, την Olaf, πώς θα ρυθμιστούν οι σχετικές διαδικασίες, όλα αυτά δεν είναι σαφή. Καλύτερα λοιπόν θα ήταν να υπήρχε ένα συνολικό σύστημα, μια συνολική διαμόρφωση του συστήματος και ιδιαίτερος καλό θα ήταν να υπήρχε σαφήνεια στην όλη αυτή τη διαδικασία. Ούτε αυτό είναι απλό βέβαια σε ό,τι αφορά και το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και σε ό,τι αφορά το Eurojust. Καλό θα ήταν λοιπόν να υπάρχει μια συνολική αντίληψη. Ευχαριστώ επόμενο ομιλητή για ένα λεπτό, κύριε Άνδρουσον. Η κυρία Άνδρουσον. Λοιπόν, επιφυλασσόμεθα όσον αφορά τη θέση μα για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, διότι δεν είχαμε ακόμα την ευκαιρία να ελέγξουμε τι λεπτομέρειε ε, του σχεδίου του κειμένου του Συμβουλίου, όπω είπαμε προηγουμένω. Καταρχήν, τα επιχειρήματα υπέρ είναι πολύ ισχυρά από τη στιγμή που υπάρχουν ε, ικανέ ρήτρε διαφύλαξη για θέματα της ανεξαρτησίας των εισαγγελέων και τα δικαιώματα των κατηγορουμένων. Εκατοντάδες εκατομμύρια, μη μπό δισεκατομμύρια ευρώ χάνονται κάθε χρόνο λόγω απατών κατά των ευρωπαϊκών ε, πόρων. Και στον Ηνωμένο Βασίλειο λυπούμε αντίθετα με αυτά που ακούσατε προηγουμένω, δεν παίρνουμε στα σοβαρά το θέμα, αρκετά σοβαρά, εάν συγκρίνουμε 38 θέματα παρεπέμφθησαν από τη Γερμανία στην, Ευρωπαϊκή, στο Ευρωπαϊκή, στην Εισαγγελία, μόνο τέσσερις στη Βρετανία. Είναι απαράδεκτο να μην έχουμε σωστή ε, ευθυγράμμιση όσον αφορά τα στοιχεία μας, τα στατιστικά για τις απάτες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η ιδέα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι καλό παράδειγμα όσον αφορά τις απάτες κατά των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάτι το οποίο είναι αναλυθές. Ευχαριστώ. Ο κ. Βοητσκόφσκι, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η ιδέα για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δείχνει ότι υπάρχει μια πολύ ανετική τάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια είναι η τάση? Όλο και λιγότερα χρήματα, αλλά όλο και περισσότερες εξασίες, όλο και λιγότερη βοήθεια και όλο και περισσότερη καταστολή. Εγώ υπενθυμίζω ότι ο προπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι λιγότερο από το 1% του ΑΕΠ και η εξουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάει προς το 100% των ελέγχων όσον αφορά τα τεκτενόμενα εντός των ευρωπαϊκών κρατών μελών. Δεν συμφωνώ με αυτές τις εξελίξεις, δεν θέλω τέτοιες ε, αλλαγές. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έπρεπε να είναι ένας θεσμός που βοηθά τους πολίτες, που ε, τίνει το χέρι προς τους ε, πολίτες και δεν οδηγείται σε αντίπεινα και σε καταστολή. Και γι' αυτό δεν θέλω να δημιουργηθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να αντικαταστήσει τις Εθνικές Εισαγγελίες. Ευχαριστώ. Επόμενος για ένα λεπτό. Yes, thank you. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε. Εγώ θέλω να σας πω ότι είμαστε υπέρ του να συγκροτηθεί αυτή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έτσι θα μπορέσουμε καλύτερα να έχουμε ε, την δίωξη της ε, διαφθορίας, διαφθοράς στην Ευρώπη που την μαστίζει. Οπότε θα πρέπει να δούμε πώς θα έχει αρμοδιότητες για τα εγκλήματα τα διασυνοριακά σε σχέση με το διεθνές δίκαιο και είναι σωστή πρώτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα πρέπει να είναι αυθεντικά ανεξάρτητη η εισαγγελία θα πρέπει να μην έχουμε προβλήματα όσον αφορά την ιστονομική συνεργασία για την τρομοκρατία και για τις ε, απάτες που φύγουν την κοινότητα. Ε, δεν θα πρέπει να έχουμε γεγονότα δυσάρεστα όπως είχαμε στην Ισπανία ε, και θα πρέπει να μην υπάρχει κανός είδους χαριστική συμπεριφορά θα πρέπει να υπάρχει ανεξαρτησία γιατί είδατε τι έγινε με, ε, με τους υπεύθυνους των χρηματοοικονομικών του Λαϊκού Κόμματος στην ε, Ισπανία. Κάτς διάει τελευταίος. Κύριος Γιαβό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτά τα ονόματα, αυτά τα συζητάμε τώρα έχουν να κάνουν με τη διαφθορά, την διασυνοριακή απάτη, την απάτη της βάρος του χρήματο Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά, ω την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, πρέπει να συμφωνήσουμε την πρόταση. Όμω, πολλά κράτη-μέλη είναι κατά τη πρόταση. Ε, φοβούνται ίσω. Φοβούνται ότι η εισαγγελία θα φέρει αυτά τα κράτη-μέλη σε ε, αμηχανία. γιατί θα έχουν κάνει απάτες αυτοί που είναι αντίστοιχοι. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχει ανεξαρτησία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έτσι θα λειτουργήσει αποτελεσματικά και όχι μόνο στα χαρτιά. Επίσης έχουμε να κάνουμε και με την αντιμετώπιση της απάτης για τον ΦΠΑ. Ε, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να ασχοληθεί και με αυτό. Χρειάζεται λοιπόν μια εισαγγελία που αυθεντικά θα είναι ανεξάρτητη και θα ασχολείται με αυτό. Και τώρα η κυρία Γιούροβα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ για τη συζήτηση. Ευχαριστώ για τη γνώμη σας που μας εξηγήσατε και για όλους ε, ε, όσοι μίλησαν υπέρ της συγκρότησης αυτής της υπηρεσίας. Θα ήθελα τώρα να δούμε το ότι είναι δική μας υψίστη προτεραιότητα και δική μου προσωπικά. Οπότε, να υπάρχει εναρμονισμένη ενιαία διαδικασία και αντιμετώπιση των εγκλημάτων κατά των οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να υπάρξουν αυτά αποτελέσματα. Οι δε φορολογούμενοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, τους αξίζει να υπάρξει ένα θεσμικό όργανο που να προστατεύει τα οικονομικά του συμφέροντα. Πιστεύουμε ότι οι απάτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση φτάνουν ε, ακόμα και τα δύο δις ετησίως. Ε, όλα αυτά θα ανακτηθούν και θα ξαναπέσουν στον προπολογισμό των, τους εθνικούς προπολογισμούς ή τον κοινοτικό. Είναι πολλά λεφτά. Πρέπει να τα εξασφαλίσουμε, να τα περιχωρήσουμε και νομίζω ότι θα πιάσουν τόπο τα χρήματα που θα δαπανίσουμε για τη λειτουργία της αγγελίας. Θα συνεργάζεται η εισαγγελία με την Όλαφ και την Eurojust. Και πολύ σωστά ελέγχθη το ότι χρειάζεται ενδελεχής προετοιμασία ενός κανονισμού που θα προβλέπει τα τη συνεργασίας αυτών των υπηρεσιών γιατί θα πρέπει η συνεργασία τους να είναι αποτελεσματική. Πολλά έχουν να γίνουν ακόμα οπότε θα πρέπει να δούμε και πώς θα υπάρξει σαφής οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων σε κεντρικό, εθνικό επίπεδο, διαφάνεια όσον αφορά το ποιοι θα αναλάβουν θέσεις εκεί Άρα προϋποθέσεις και κριτήρια να είναι αυστηρά, ανεξαρτησία, αμεροληψία, επαγγελματισμό όσων θα επιλεγούν. Επίσης, σωστά ελέγχθη ότι τα δικονομικά δικαιώματα δεν θα πρέπει να θυσιάζονται. Θα πρέπει να είναι κατοχυρωμένα και στα πλαίσια των ενεργειών της ε, εισαγγελίες. Έχουμε τώρα αυτές τις κίτρινες κάρτες που προέρχονται από πολλά κράτη-μέλη και από τα κοινοβουλιά τους. Ε, δεν θεωρώ ότι αυτά έβαλαν τα φόπλακα στην πρόταση. Κάποια κοινοβούλια. Ε, ήρθαν σε επαφή μαζί μου, ε, έγιναν και κάποιες επισκέψεις τους εξήγησα ότι υπάρχουν ασφαλιστικές δικλίδες. Δεν θα παραβιάσουμε την επικουρικότητα. Δεν θα μπούμε στα χωράφια τους, δεν μπούμε στα χωράφια των εθνικών δικαστηρίων. Οι αρμοδιότητες των εθνικών δικαστηρίων θα διατηρηθούν. Αυτά τους είπα και πολλά άλλα. Και νομίζω ότι τελικά διατίθενται φετικά αυτά τα κοινοβουλία μπορέσαμε με αυτή την επικοινωνία να καταλήξουμε στο ότι δεν θα υπάρξει παραβίαση της αρχής της επικουρικότητας. Και πάλι ευχαριστώ κύριε και κύριοι. Παρακαλώ αύριο στην ψηφοφορία να επιψηφίσετε την πρόταση για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ευχαριστώ και στο τέλος η κυρία Μακοβέη, η συγκητριά μας έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η συζήτηση ήταν άκρος ενδιαφέρουσα. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε κάποιες τεθήσεις ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα, ρητορική ερώτηση που απευθύνεται προς τους συναδέλφους των κρατών μελών εκείνων που είναι κατά ή που ανήκουν σε πολιτικές ομάδες που είναι κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Λοιπόν, που από τις δικές σας έρευνες στη δική σας χώρα πόσα χρήματα ανακτήθηκαν από τους ευρωπαϊκούς πόρους που εκλάπησαν. Λίγα, πολλά, μεγάλα ποσά, μικρά ποσά. Ίσως δεν θέλουν να φαίνεται το έργο της Εθνικής Αγγελίας. Ε, δεύτερη ερώτηση, σημαντικότατη. Το χρήμα των φορολογουμένων μας. Βρίσκεστε σε ένα κοινό κορβάνα. Όλα αυτά τα χρήματα λοιπόν όσο βρίσκονται εκεί στον ίδιο κορβανά θα πρέπει να τα προστατεύουμε όλοι. Αν σε μια χώρα τα πράγματα πηγαίνουν πολύ καλά και οι έρευνες διενεργούνται και ολοκληρώνονται και δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο σε άλλη χώρα, αυτό σημαίνει ότι κλέβουμε χρήματα και από τους πολίτες των χωρών όπου τα πράγματα λειτουργούν καλά. Τώρα, για τους συναδέλφους των κάτω χωρών που αναφέρθηκαν ότι στην πατρίδα τους οι έρευνε πραγματοποιούνται καλά. Ναι, αλλά σε άλλε χώρες δεν ισχύει κάτι τέτοιο και τα χρήματα είναι σε κοινό κορβάνα. Λοιπόν, τρίτον, η ανεξαρτησία των εισαγγελέων έναντι το, του πολιτικού τομέα. Πιστεύω ότι ο κύριος Νεγκρέσκου μίλησε λέγοντας ότι θέλει αυτή την ανεξαρτησία και ότι τώρα στη Ρουμανία στο ρουμανικό κοινοβούλιο ε, θεωρούνται από διαφορετική οπτική γωνία. Έχουν διαφορετική άποψη στο Ρουμανικό Κοινοβούλιο. Είναι προφανές ότι και για τους εισαγγελεί των κρατών μελών και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πρέπει να επικρατεί μια ανεξαρτησία. Τέταρτον, θέλουμε επίσης να διώκονται και οι παραβιάσεις κατά του, οι παραβάσεις που στρέφονται κατά του ΦΠΑ. Πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι για να μειωθούν οι απάτες κατά των ε, ευρωπαϊκών συμφερόντων. Ευχαριστώ συνάδελφοι. για αυτή τη συζήτηση. Πρέπει πάμε στο επόμενο σημείο της ημέρης διάταξης.